the president Good afternoon, colleagues. The session... Ε, καλησπέρα σας συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η σύνεδρος που διακόπησε στις 16 του μηνός. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η Ολομέλεια. Καθίστε παρακαλώ.